Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ. Παρακαλώ. Ας ξεκινήσουμε αυτή την κοινή συνεδρίαση Econ και Budget. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Προπολογισμού, Ζαν Αρτουή, ε, ζητά συγγνώμη που δεν μπορεί να είναι εδώ, αλλά παρακολουθεί μια άλλη συνεδρίαση με την Επιτροπή για την αναθεώρηση του, του δημοσιονομικού πλαισίου, αλλά θα συμπροεδρεύσω με τον κύριο Μούρεσαν, Πρόκειται για κοινή συνεδρίαση που είναι αφιερωμένη στην έκθεση για την ε, δημοσιονομικές δυνατότητες της Ευρωζώνης. Είναι μια έκθεση προόδου μετά από την τελευταία κοινή συνεδρίαση που είχαμε στις 12 Ιουλίου. Ε, να σας θυμίσω ότι Υπάρχει ισχυρή πολιτική βούληση για να κλείσει η έκθεση αυτή πριν το τέλος του έτους, να υιοθετηθεί μαζί με τις ε, δύο εκθέσεις της ΑΦΚΟ για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί τη βάση του δυναμικού της συνθήκης του Λισαβόνας καθώς και τις πιθανές εξελίξεις και προσαρμογές του σημερινού θεσμικού πλαισίου. Να σας πω από την συνεδρίαση των σκιωδών που έγιναν μάλλον οι εισηγητές θα μας ενημερώσουν για τις ε, συνεδριάσεις των ε, σκιωδών και θα μας ε, πούν επίσης που βρισκόμαστε και χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση δίνω το λόγο στον κύριο Μπέγκε. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ευχαριστώ που είστε εδώ παρά την προκεχωρημένη ώρα. Είχαμε δύσκολες ζητησεις και συνεδριάσεις και με τους κοιόδης ηγητές από τις ομάδες Πάντα υπάρχουν φάσεις δύσκολες σε αυτά τα θέματα. Πρέπει να μελετήσουμε περισσότερα τα θέματα λοιπόν επί τη βάση αυτών των συζητήσεων. Ως έχουμε ετοιμάσει ένα έγγραφο το οποίο πιστεύουμε ότι μπορεί να δώσει καθοδήγηση για να προχωρήσουμε και να συμφωνήσουμε ως πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο. Μια τέτοια έκθεση βέβαια πρωτοβουλία αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να επισέλθει σε λεπτομέρειες νομοθετικές. Δεν πρόκειται καν για έκθεση μίας μόνης ομάδας. Είναι ένα έγγραφο κοινό και ω εκ τούτου περιλαμβάνει συμβασμούς και μάλιστα δύσκολους. Θέλω εκ προημίου να επισημάνω ότι όταν αναφερόμαστε και σε διάφορες εκθέσει των τεσσάρων ή πέντε προέδρων λόγος, ε, έχουμε πρώτα απ' όλα το Διεθνέ Οσμοτικό Ταμείο, το οποίο από πέρσι, αλλά επανειλημμένω, έχει ζητήσει ε, μέσα τα οποία θα λειτουργούν καλύτερα, έχει παρουσιάσει μέτρα τα οποία θα λειτουργούν καλύτερα και στο βαθμό που δεν τα έχει καλύψει επαρκώς τον εγγραφό μας, παρακαλούμε να συμπληρώσετε εσείς. Το ζήτημα λοιπόν ε, των δυνατοτήτων και των ε, προϋποθέσεων θα έχει πολύ σημαντικό ρόλο στην υπόθεση αυτή. Δηλαδή, δεν έχουμε επιτύχει αυτά που θα θέλαμε, ξεκινώντας ε, τη λειτουργία του ευρώ και οι παρεμβάσεις με το 4-pack, το 6-pack κτλ. Ε, δεν πρέπει βέβαια να θεωρηθούν αμελητές, αλλά πρέπει να εξετάσουμε παρόλα αυτά τι συμβαίνει τι θα κάνουμε, πώς μπορούμε να προετοιμαστούμε και τι διδάγματα έχουμε να αποκομίσουμε εν ώψη προηγούμενων κρίσεων και ενδεχόμενων μελλοντικών, γιατί θα υπάρξουν και στο μέλλον κρίσεις. Σε αυτό προσπαθήσαμε λοιπόν να τοποθετηθούμε. Έχουμε ένα φύλλο πορείας συντάξει με βάση και τα πρώτα έγγραφα εργασίας για τις προτάσεις και ενσωματώνοντας βέβαια πάντα τις τροπολογίες πνεύμα συμβασμού για να έχουμε ένα σύντομο, ευανάγνωστο και σαφές ως προς την καθοδήγησή τους προς προσανατολισμούς του έγγραφου. Προσπαθούμε λοιπόν και να καταγράψουμε την κατάσταση όπως έχει τώρα και να εκθέσουμε γενικές αρχές οι οποίες από ό,τι βλέπω τουλάχιστον την χάνουν γενικής αποδοχής από τις συζητήσεις με τους και ηγητές, τουλάχιστον αυτό βλέπω. Και στο κεφάλαιο που αφορά εμένα περισσότερο, τους τρεις πυλώνες, το fiscal capacity, τη σύγκληση, τη σταθεροποίηση της Ευρωζώνης, έχουμε κάνει αυτή την κατανομή. Έχουμε ακόμη ένα κομμάτι που αφορά τη διακυβέρνηση, δημοκρατική λογοδοσία και έλεγχο. Και έχουμε συζητήσει με τους συναδέλφους όλα αυτά τα θέματα για να ανοίξουμε στη συνέχεια το δρόμο για ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές και επί τη βάση βέβαια των προτάσεων που θα καταθέσουμε εδώ ε, και για τη Ρωμή 4. Ένα πλαίσιο για μακροπρόθεσμη σταθεροποίηση της Ευρωζώνης. Και ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια λευκή βίβλο με ένα φιλόδοξο κεφάλαιο και για την Ευρωζώνη και, για τις νομοθετικές προτάσεις που θα πρέπει να κατοτεθούν μέσα στο 2017. Θα αξιοποιήσουμε κάθε δυνατότητα βέβαια για συνεννόηση πέραν των κομματικών γραμμών για να προτείνουμε και νομοθετικά μέτρα και να ανοίξουμε το δρόμο μέσω και μακροπρόθεσμα για όποιες απαραίτητες ε, ε, τροποποίησεις και στις συνθήκες. Νομίζω ότι με το έγγραφο αυτό έχουμε μία βάση που μπορεί να προχωρήσει, μπορεί να γίνει αποδεκτή ευρύτερα. Βεβαίω θα πρέπει να συζητήσουμε τα επιμέρου σημεία. Έχουμε βρει έναν δρόμο, αλλά πρέπει να δούμε και σε σχέση με άλλα κύματα πώ μπορούμε να διαμορφώσουμε συμβαστικέ λύσει. Είμαστε βέβαια δεκτικοί σε κάθε πρόταση και θα αξιολογηθούν όλες οι προτάσεις και μέσα στις ομάδες μας ασφαλώς. Και νομίζω κύριε Πρόεδρο, Πρόεδρε ότι πρέπει να τηρήσουμε πάνω απ' όλα το χρονοδιαγραμμό, ώστε να πάει το κείμενο με την έκθεση στην Ολομέλεια το Δεκέμβριο. Έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τις θέσεις μας εν ώψη ε, και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου και να είμαστε έτοιμοι για τη Ρώμη το Μάρτιο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, και για τις αφείς θέσεις ε, και την έκθεση του χρονοδιαγράμματος. Κύριε Μπερές. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καθώς πρόκειται για ε, κοινή έκθεση και σήμερα παρουσιάζουμε το φύλλο πορείας ε, από το, οποίο υπάρχει σχεδόν πλήρης συνένεση ανάμεσα στους συνεισηγητές. Δεν έχω πολλά να προσθέσω. Θα ήθελα απλά να πω δύο λόγια για τη μέθοδο, διότι το φύλλο αυτό πορείας που σας παρουσιάζουμε, ορισμένοι θα το βρουν πολύ σύντομο και άλλοι θα χαρούν για την σαφήνεια του μηνύματος. Και ίσως ε, επειδή έχουμε περάσει πολλά χρόνια στο Ευρωκοινοβούλιο, οι δύο συνεισηγητές θελήσαμε να βγούμε από τη λογική σύμφωνα με την οποία επειδή θέλουμε όλους ε, να τους ε, έχουμε ικανοποιημένους να κάνουμε διάφορες φράσεις ε, συνεννόησης όπου δεν φαίνεται τι, ποια είναι η ουσία. Θελήσαμε να έχουμε ένα σαφές μήνυμα, ένα πολιτικό μήνυμα όπου στη, τη στιγμή που καθένας ε, βλέπει ότι το ευρώ δεν μπορεί να σταθεί μακροχρόνια χωρίς ουσιαστικές ε, αλλαγές και μετά από τον Brexit θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να σταθεροποιήσουμε και να παγιώσουμε το ευρώ ως δομικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκή Ένωση, πιστέψαμε ότι το, ο ρόλος του Ευρωκοινοβουλίου ήταν να στείλει μήνυμα πολιτικό, σύντομο και σαφές. Μέσα σε αυτό το πνεύμα δουλέψαμε και ξανά δουλέψαμε για να καταλήξουμε σε αυτό το φύλλο πορείας. Υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο προτείνεται το Φιλοπορίες, όπου τίθεται βεβαίως το θέμα του Brexit και που έχει πολύ μεγάλο αντίκτυπο στο πνεύμα που επικρατεί στη συζήτηση πριν καν ανατεθεί επιτάπητος το άρθρο 50 στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Και ο κίνδυνος που ελοχεύει είναι ότι κάθε συζήτηση που έχει να κάνει με την Ευρωζώνη να είναι ένα θέμα διχασμού για τους 27 αυτό το, επίσης δεν το πιστεύουμε οι δύο συνεισηγητές. Πιστεύουμε ότι όποιο και αν είναι το κοινό θέμα γενικού συμφέροντος, τα όσα αφορούν την Ευρωζώνη δεν μπορούν να περάσουν σιωπηρά. Και γι' αυτό είναι σημαντικό όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει το λευκό της βιβλίο, η εντολή διευρύθηκε στην Πρατισλάβα για ένα σύνολο, συνολικό όραμα για τους 27 ε, αυτό το θέμα να μην περάσει σιωπηρά. Και δύο τελευταίες παρατηρήσεις. Η πρώτη είναι ότι προφανώς ορισμένες από τις προτάσεις που υποβάλλουμε θα χρειαστεί να οδηγήσουν σε αναθεώρηση της συνθήκης. Ε, όμως δεν θελήσαμε να οργανώσουμε τη σκέψη μας μόνο και μόνο με βάση αυτό το κριτήριο. Γιατί ξέρουμε ότι τόσο η Επιτροπή του Προπολογισμού όπως και η Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή, ρόλος μας δεν είναι καταρχάς πώς θα οργανώσουμε την εφαρμογή της τάδε δίνα πρότασης, αλλά να υποβάλουμε προτάσεις. Ποιες είναι οι προτάσεις που πρέπει να υποβληθούν ώστε το ευρώ να μπορεί να σταθεί ε, ε, βιώσιμα. Έπειτα έχουμε και το θέμα του χρονοδιαγράμματος που είναι σημαντικό γιατί γνωρίζουμε ότι και άλλε εκθέσεις συντάσσονται στο Ευρωκοινοβούλιο ιδιαίτερα όσον αφορά την, ε, το κύριο, ε, μάλλον υπό την ε, Συνταγματική Επιτροπή που θα πρέπει να εγκριθούν ταυτόχρονα με είναι εδώ ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να είναι σε θέση να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα στο, στο Συμβούλιο και στην Κομισιόν. Ευχαριστώ. Κύριε Μούρεσαν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Εξ ονόματος ε, των ε, συναδέλφων του ΕΛΚ στην ε, ΕΚΟΝ θα πρέπει να σας πω ότι στη διάρκεια του έτους είχαμε διάφορες σκέψεις και σε επίπεδο σκιωδών εισηγητών. Θέλω να ευχαριστήσω τους δύο συνεισηγητές για την εργασία και την υπομονή με την οποία δούλεψαν στη διάρκεια του έτους. Βεβαίως πρόκειται για δύσκολο θέμα και αυτό μπορούμε να το αναγνωρίσουμε μόνο και μόνο από το γεγονός ότι πάνω από 800 τροπολογίες υποβλήθηκαν από συναδέλφους ε, από τις διάφορες ομάδες. Τώρα που βρισκόμαστε. Έχουμε μία εκδοχή της έκθεσης υπό τη μορφή φίλου πορείας ε, που βεβαίως σας έχει σταλεί νωρίτερα σήμερα και επί τις οποίες μέσα στο ΕΛΚ, στην ομάδα της ΕΚΟΝ, θα πρέπει να διαβουλευτούμε και να δούμε σε ποιο βαθμό οι κόκκινε γραμμέ που έχουν εκφράσει οι συνάδελφοι τηρούνται εδώ και περιλαμβάνονται εδώ. Ποια είναι η θέση του ΕΛΚ στην ΕΚΟΝ και ποιε ήταν οι κόκκινε γραμμέ. Είπαμε εξ αρχή ότι θέλουμε να παίξουμε επικοδομητικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία και αυτή τη συζήτηση. Θέλουμε να προγραμματιστούμε για τον όγκο τη δημοσιονομική ε, δυνατότητα, πόσο θα πρέπει να σωρεύσει αυτή η ε, δυνατότητα και από πού θα προέλθουν αυτά τα χρήματα και τι θα πρέπει να χρηματοδοτήσει. Και όσον αφορά τον όγκο, βεβαίως πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Αν πάμε στα κράτη-μέλη, και που του ζητήσουμε ε, άμεση συμβολή σε μια ε, δημοσιονομική δυνατότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πόσο έτοιμοι θα είναι να συμβάλλουν με άμεσες πληρωμές. Στοχεύουμε για έναν ίδιο πόρο μέσω και μακροπρόθεσμα. Ε, αυτή θα ήταν η προτιμότερη εκδοχή, αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε και τρόπους για να το εφαρμόσουμε αυτό και να αξιολογήσουμε ποιοι και κατά πόσο ήδη οι πόροι είναι εφικτοί μέσω και μακροπρόθεσμα. Επίσης αναφέρεται στο ε, φιλοπορίες ότι αυτός, αυτή η δυνατότητα θα, πρέπει να μπορεί να διασώσει ένα μεγάλο κράτος μέλος που βρίσκει δυσκολίες και χρειάζεται 500 με 1000 δις. Δηλαδή ένα τρεις. Από πού θα έρθουν αυτά τα χρήματα. Και επίσης θα πρέπει να σκεφτούμε ότι αυτή η δυνατότητα δεν θα πληρεί την ίδια λειτουργία όπως ο ESM γιατί Υπάρχει ήδη αυτός, άρα λοιπόν θα πρέπει να είναι ρεαλιστικό σε όγκο μια τέτοια δυνατότητα. Θα πρέπει να εμποδίζει τις χώρες να μπουν σε κρίση, να, να, να δίνει κίνητρα για μεταρρυθμίσεις και αν πάρει τη μορφή ενός κονδυλίου ε, για, το, για χαλεπούς καιρούς, ε, θα πρέπει να, υπάρχει, να υπάρχουν διαφορετικές δυνατότητες. Μια από τις γραμμές που είναι στο φύλλο πορείας και προήλθε από το ΕΛΚ και αυτό ήταν και θέμα ανοιχτή συζήτηση, είναι το σχέδιο για ε, επίδομα ανεργίας. Οι συνάδελφοι του ΕΛΚ το απορρίπτουν μέχρι στιγμής και αυτό δεν θα αλλάξει μια πρόταση και είναι τα τελευταία που θα πω Πρόεδρε, μια επιπλέον πρόταση που αναφέρεται στο φύλλο πορεία είναι ο υπουργό Οικονομίας. Εδώ ε, Λέμε ότι έχουμε δημοσιονομικούς κανόνες στην Ευρώπη και η προτεραιότητα θα πρέπει να είναι ο σεβασμός και η εφαρμογή τους. Μιλάμε για το διπλό πακέτο, για το εξαπλό πακέτο, για το οποίο υπήρχε σαφής πλειοψηφία στην περασμένη θητεία εδώ και η αντίληψή μας είναι ότι αυτοί οι κανόνες υπάρχουν και πρέπει να εφαρμόζονται αυτόματα. Για όλα τα κρατημέλη με τον ίδιο τρόπο. Και ότι δεν θα πρέπει άλλο να νερωθούν αυτοί οι κανόνες. Και ο στόχος για την ύπαρξη ενό Υπουργού Οικονομίας θα ήταν να, μπορεί να εφαρμόσει και να ενσωματώσει τους κανόνες αυτούς στην Ευρώπη. Και ε, εδώ έχουμε μεγάλες δυσκολίες από την πλευρά του ΕΛΚ. Τα τονίζω γιατί είναι σημεία που πρέπει να δουλέψουμε ακόμα. Κατά τα άλλα, νομίζω πως έχει σημειωθεί εξωσημείωτη πρόοδο τους τελευταίους μήνες και υπήρχε σαφής βούληση από πλευρά της ομάδας του ΕΛΚΑ στην ΕΚΟΝ να υπάρξει αυτή η πρόοδο. Σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ γιατί μιλήσατε για τη δημοσιονομική ικανότητα. και παρουσιάσατε το λογικό επιχείρημα. Επόμενος ομιλητής, ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω τους εισηγητές και τους ισκιώδες εισηγητές που δυσκολεύουν τη συζήτηση ενίοτε, αλλά την κάνουν και πιο επικοδομητική. Νομίζω ότι έχουμε ένα φιλοπορία σε αυτό το νοδικό χάρτη. Είναι μια πολύ καλή κίνηση αυτή, γιατί δίνει ένα σαφές πολιτικό μήνυμα και αυτό είναι σημαντικό για το Κοινοβούλιο, να δείξει ότι το ευρώ δεν είναι βιώσιμο έτσι όπως έχει αυτή τη στιγμή και πρέπει να το καταστήσουμε βιώσιμο. Και για να μπορέσει και θα πρέπει να κάνουμε τα πάντα έτσι ώστε το ευρώ να λειτουργήσει προς όφελος των κρατών μελών και των λαών. Να το κάνουμε λοιπόν να λειτουργήσει. Αυτό είναι το σημαντικό. Είναι ένα σημαντικό μήνυμα που πρέπει να ακουστεί χειρά και αυτό το φιλοπορία δείχνει ε, ποιες λειτουργίες του συστήματος πρέπει να ρυθμιστούν και να εξεταστούν καλύτερα για να γίνει το ευρώ βιώσιμο. Και καλώς. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι εδώ πρέπει να διαχωρίσουμε ξεκάθαρα τις εθνικές από τις ευρωπαϊκές αρμοδιότητες. Εάν πρόκειται να έχουμε ένα σύστημα διακυβέρνησης θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ποιος έχει αρμοδιότητα για ποιο πράγμα. Και σε αυτή την περίπτωση βλέπουμε ότι λειτουργούμε υπό δυσχερείς συνθήκες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν φαίνεται σαν κάτι το καλό, αντίθετα δίνει την εικόνα της απειλής και του κινδύνου ενίοτε και πρέπει να δείξουμε ότι δεν είναι μια ένωση που θα επεκτείνεται και θα διαστέλλεται στο άπειρο, ότι αυτή η πρόταση συμφέρει όλους και θέλει να κάνει το ευρώ να λειτουργήσει σωστά για όλους. Και πιστεύω ότι αυτός ο διαχωρισμός μεταξύ των ε, εθνικών αρμοδιοτήτων και των ευρωπαϊκών αρμοδιοτήτων είναι θολός και δεν είναι καλό αυτό το πράγμα. Ε, με δυσαρέσκεια διαπιστώνω ότι οι ιδιώτες επενδυτές μπορούν να επηρεάσουν κάποιο, κάποια νομοθετική διαδικασία πολύ περισσότερο ίσως από τους φορολογούμενους στο παρελθόν. Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται η ιδιοκτησία από τα κράτη-μέλη. Δεν είναι μόνο δουλειά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα πρέπει οι εθνικοί πολιτικοί, άνδρες και γυναίκες στην εκάστοτε χώρα να έχουν την ιδιοκτησία ε, αυτού του εγχειρήματος. Και χαίρομαι διότι μου δίνει την ευκαιρία να το υπογραμμίσω για άλλη μια φορά. Νομίζω ότι είμαστε σε καλή στιγμή και ότι θα τηρήσουμε τα χρονοδιαγράμματα χωρίς πρόβλημα. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ο κύριος Λούκε για τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές. Ο κύριος Χου... Η κυρία Πέτρα Χουγκόνεν. Ρούοχόνεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφους ε, για την προσπάθειά τους να βρουν μια διέξοδο στην υπόθεση αυτή. Αλλά πρέπει να πω ότι αυτό το φιλοπορία δεν με πείθει ότι είναι αναγκαία η προσέγγιση που προτείνει. Έχω άλλωστε κάνει σχετικά σχόλια και στο παρελθόν. Το Ταμείο για τα Απρόβλεπτα δεν νομίζω ότι μπορεί να περιορίσει τον λεγόμενο ηθικό κίνδυνο moral hazard. Για μένα δεν αρκεί και δεν, είναι, δεν αρκεί η εστίαση στον ε, ηθικό κίνδυνο και δεν νομίζω ότι το ε, Ταμείο για τα Απρόβλεπτα θα μπορούσε να δώσει απαντήσεις σε προβλήματα αντίστοιχα με αυτά της ελληνικής κρίσης εάν εμφανίζονταν στο μέλλον. Κάτι ακόμη. Ένα γενικό πρόβλημα είναι η περιστολή της εθνικής κυριαρχίας στην υπόθεση αυτή, όπως διαγράφεται. Δεν θα είμαι σε θέση λοιπόν να υπερασπιστώ έναντι του ψηφοφόρου μου αυτές τις προτάσεις. Νομίζω ότι πρέπει να εστιαστούμε περισσότερο στο να καταστήσουμε πιο αποτελεσματικό και πιο απλό το ισχύον σύστημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριο Κέλμερ είναι εγγεγραμμένο στο κατάλογο των ομιλητών, αλλά παίρνετε εσεί το λόγο εκ μέρου του. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εκπρόσωπο τον κύριο Κέμελ, κύριο Λούκα. Πολύ σύντομα, δεν ξέρω αν έχω διαβάσει το ίδιο έγγραφο με αυτό που μα σχολίασαν οι συνάδελφοι, Μπόγκοσταν και άλλοι, γιατί δεν διαπιστώνω καμία πρόοδο, ούτε ευόδοση χάρη στο έγγραφο αυτό των προσπαθειών μας. Υπάρχουν ε, μεγάλα χωρία του εγγράφου, τα οποία απλώ δεν θέση να αντιληφθώ. Αλλά ίσως αυτό έχει να κάνει και με τις περιορισμένες μου δυνατότητε κατανόησης των εγγράφων σε σχέση με άλλου συναδέλφους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Νομίζω ότι υπάρχει μια εικόνα, μια καταγραφή της πολιτικής, του πολιτικού κλίματος εδώ και της οικονομικής κατάστασης. Επομένως, ε, δεν ξέρω αν είμαι σε θέση να το δεχθώ. Σας ευχαριστώ. Ο Φάμπιο Ντεμάση. Oh, sorry, sorry, sorry. Με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε, ζητώ συγγνώμη. Λόγω κούρασης. Ο κύριος Στόρβαλτς. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω τους εισηγητές Είχαμε διασκεδαστικές στιγμές και κάποιες λιγότερο διασκεδαστικές κατά τη σύνταξη αυτή, αυτού του κειμένου. Ενίοτε η συζήτηση ήταν σαν να ήταν μια εικονογράφηση για το βιβλίο «Το ευρώ και η μάχη των ιδεών». Ξέρετε, σε στιγμές κρίσης όλοι θέλουν τους πολύ ισχυρούς κανόνες. Και στη συνέχεια αρχίζει η συζήτηση για το πώς θα παρακαμφθούν οι κανόνες. Και αυτό κυριάρχησε στις συζητήσεις μεταξύ των σκιωδών εισηγητών. Οφείλω να σας πω. Τρία είναι τα βασικά σχόλιά μου για το κείμενο, έτσι όπως έχει αυτή τη στιγμή. Πρώτον, με δυσαρεστεί το γεγονός ότι αποδυναμώθηκε το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, η διατύπωσή του με το διπλό και το εξαπλό πακέτο, Το λέω αυτό και σε σχέση με αυτά που είπε ο συνάδελφος ο κ. Μόρισαν. Μετά έχουμε το δεύτερο πυλώνα και την αυτόματη παρατήρηση, αν θέλετε, της εκάστοτε κρίσης θα πρέπει να βάλουμε μια τελεία πριν μπούμε στις λεπτομέρειες. Αυτό είπαμε στη συνάντηση των σκιωδών εισηγητών. Θα μπορούσα ενδεχομένω να δεχθώ το Ταμείο για τα απρόβλεπτα και ίσως να μπορούσαμε να καταλήξουμε σε σωστούς κανόνες για τον τρόπο με τον οποίο θα το διαχειριζόμαστε Όμω πάντοτε φοβάμαι ότι θα υπάρχουν τζαμπατζίδε εάν, εάν πραγματικά υπάρξει αυτό το ευρωπαϊκό καθεστώς ε, επιδόματος Ανεργία Αυτό το δεύτερο ε, πρόγραμμα για την ενίσχυση των αναέργων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί ξέρετε, αυτά τα προγράμματα δεν δόθηκαν σαν ε, πρωινό δώρο στον καθένα που θέλει να είναι τζαμπατζής, αλλά φτιάχτηκαν από τα συνδικάτα. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε εδώ πολύ συνεκτικοί και συνοπτικοί στη διατύπωση και να μην βγούμε σε λεπτομέρειες. Και η τρίτη παρατήρηση που έχω να κάνω, την έχω ήδη αναφέρω, αναφέρει. Ξέρετε, υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα παράθεση των λόγων κάποιου. Feeding investment reach full employment aggregate demand. Το διάβασα αυτό και φαντάστηκα ότι είναι πλήρης αντιγραφή του βιβλίου του σχετικού του John Maynard Keynes, το οποίο δημοσιεύτηκε το 1936, όπου το βάρος του δημοσίου χρέους ήταν εξαιρετικά μικρό. Συγκριτικά με αυτό που έχουμε τώρα. Ότι δηλαδή οι μεγάλες επενδύσεις θα οδηγήσουν αθρηστικά στην αύξηση της ζήτησης. Κάτι το οποίο είναι καλό για την οικονομία. Νομίζω ότι θα πρέπει να μην είμαστε τόσο πολύ ένθερμοι οπαδοί και υποστηρικτές του εκέινσιανισμού και να μην παραθέτουμε τσιτάτα του 1936. Σε κάθε περίπτωση ο μιλωτής που μίλησε για την ιδιοκτησία, την εθνική ιδιοκτησία ε, των αποφάσεων ε, έχει απόλυτο δίκιο. Και αυτό μένει να δούμε και μπροστά μας. Αυτό έχουμε μπροστά μας στο μέλλον. Πρέπει να γίνει μια πραγματική πραγματικά ειλικρινής και σε βάθος συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο τα εθνικά κράτη και τα εθνικά κοινοβούλια θα αναλάβουν το μέρος που τους αναλογεί στην ιδιοκτησία όλων αυτών των προγραμμάτων που είναι προς όφελος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Για το Άλντε θέλει κάποιος το λόγο ο κύριος Ντεμάση. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εισηγητές και να αξιοποιήσω αυτή την ευκαιρία για να διαφωνήσω με τον προηγούμενο μιλητή για το τι θα μας συμβούλευε ο Τζον Μέιναρτ Κέινς, γιατί έγραψε και ένα άρθρο για τις οικονομικές ευκαιρίες ε, των εγγονών μας. Και εκεί κατέστησε σαφές το ότι το ζήτημα των δημοσίων επενδύσεων θα αποκτούσε όλο και μεγαλύτερη σημασία με την πάροδο του χρόνου και αυτό ακριβώς παρατηρούμε μια πολύ κεινσιανή κατάσταση όπου η απόπειρα, η προσπάθεια να μειωθεί το δημόσιο χρέος με τις επιθετικές πολιτικές λιτότητας έχει αποτύχει κατά κράτο και αυτό είναι το μεγάλο παράδοξο και βεβαίως μπορούμε να το συζητήσουμε ε, γύρω από ε, δύο φλιτζάνια καφέ σε ένα πιο κατάλληλο για συζητήσεις μέρος, όμως η δημοσιονομική ικανότητα δεν είναι ένα τεχνικό εγχείρημα. Αυτό το οποίο είδαμε αυτή την εποχή και κυρίως σήμερα με την έκβαση των Αμερικανικών εκλογών είναι το ότι οι κοινωνίες πιέζονται πάρα πολύ από τις πολιτικές που εφαρμόζονται μετά το ξέσπασμα της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης. Και μόνο το σεβασμό που σας τρέφω και παρά το πολύ δύσκολο έργο σας είμαστε πολύ μακριά από συμβαστική λύση εδώ διότι διαφωνούμε θεμελιωδώς με πολλά από αυτά που λέτε. Δεν χρειαζόμαστε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που κατακρεουργούν τη ζήτηση. Δεν έχω τίποτα εναντίον των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, αλλά επιτέλους να δώσουμε ένα νόημα σε αυτή τη λέξη. Τι είδους διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις χρειαζόμαστε και δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που έχουν εφαρμοστεί τα τελευταία χρόνια, οι οποίες το μόνο που κάνουν είναι να μειώνουν δραστικά την αγοραστική δύναμη και την αθρηστική ζήτηση. Θα πρέπει να χρηματοδοτούνται τα ελλείμματα εγχωρίως με την ιδιωτική αποταμίευση και θα πρέπει να υπάρχει διόρθωση της μακροοικονομικής ανισορροπίας. Θα πρέπει να ακολουθηθεί σχετική διαδικασία και Στη δική μου χώρα, για παράδειγμα, υπάρχει υπέρβαση των πλεονασμάτων έτσι όπως έχουν οριστεί τα πλεονάσματα και τα ελλείμματα και δεν γίνεται τίποτα γι' αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε μια πλήρως ισορροπημένη και συμμετρική ε, μακροοικονομική διαδικασία και όχι να ασχολούμαστε μόνο με τα ελλείμματα και όχι τα πλεονάσματα. Και τέλος, αναφέρθηκε η ανάγκη για επενδύσεις. Και πιστεύουμε ότι το ΕΦΣΥ, το σχέδιο Juncker δεν έχει δώσει τα απαραίτητα αποτελέσματα, έχει αποτύχει δεν ε, λειτουργήσε με προσθετικότητα, θα πρέπει να ξανασυζητήσουμε τις δημόσιες επενδύσεις, να επενδύσει το κράτος πάλι. Ε, μπορούμε να ζητήσουμε και να συζητήσουμε για τα αντισταθμίσματα, τα ανταλλάγματα. Κάποιοι λένε για το επίδομα ενεργεία, κάποιοι λένε για την απελευθέρωση, πιο έντονη απελευθέρωση της αγοράς εργασίας. Ε, κάποιοι λένε για μεγαλύτερη μετακίνηση του, του, εργατικού δυναμικού. Εμείς δεν νομίζουμε ότι είναι αυτές οι βιώσιμες λύσεις. Αντίθετα, πρέπει να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης και ανάπτυξη και κυρίως στις οικονομίες της περιφέρειας της Ευρωζώνης. Και είναι εξαιρετική ευκαιρία ε, να το συζητήσουμε αυτό την επόμενη εβδομάδα της ανεπάρκειας του ευρωσυστήματος με τον Τζόσεφ Στίγκλιτς, ο οποίος θα επισκεφθεί ε, τις Βρυξέλλες την επόμενη εβδομάδα και ελπίζω να μας εμπενεύσει γιατί θα είναι ένα εξαιρετικό βήμα προς τα ε, εμπρός. Αυτά είχα να πω. Το υπόλοιπα θα το πω με τον Νίλς τέτα τέτ ε, πίνοντας καφέ κάπου αλλού. Ευχαριστώ. Δεν είναι εδώ και γι' αυτό και μίλησα λίγο παραπάνω. Μαραβάλλω. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να μιλήσω στα ισπανικά. Εγώ νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε σήμερα στο εξής. Αν δεν είχαμε ξεκινήσει αυτή τη δουλειά και ευτυχώς το κάναμε πριν από κάποιους μήνα, μήνες, σήμερα θα βλέπαμε τα αποτελέσματα των Αμερικανών εκλογών και θα λέγαμε να ένας παραπάνω λόγος επιγόντως να ασχοληθούμε με την Ευρωζώνη που μας ανησυχεί και που αποτελεί καθήκον μας. Γι' αυτό και σήμερα πρέπει να ευχαριστήσουμε τους εισηγητές για τη δουλειά τους, αλλά να αξιολογήσουμε θετικά τη στάση τους επίσης, γιατί μας επέτρεψαν να έχουμε θετική έκβαση και να υπάρχει μια επαρκή συμφωνία. Ξεκινήσαμε με πολύ μεγάλη φιλοδοξία με το πρώτο κείμενο, υπερβολική ίσως φιλοδοξία και υπήρχαν πάρα πολλές ε, τροπολογίες και καταλήξαμε σε ένα πολύ σύντομο κείμενο αλλά με μεγαλύτερες ε, πολιτικές φιλοδοξίες και ε, πιστεύουμε ότι θα είναι πολύ πιο αποτελεσματικό και πολύ πιο λειτουργικό. Το έχουμε έτσι ώστε και η Επιτροπή και το Συμβούλιο να μας το επιστρέψουν με την μορφή των νομοθετικών προτάσεων που θα ενσαρκώνουν ακριβώς τις έννοιες και τις ιδέες που έχουμε βάλει εμείς σε αυτό το σύντομο κείμενο. Έχουμε ξεκάθαρα εκφράσει τη στάση μας, θέλουμε να συνεργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση, να είμαστε αποτελεσματικοί για να καλύψουμε τα κενά και την ε, ανεπάρκεια της Ευρωζώνης, την οποία όλοι γνωρίζουμε και όλοι αποδεχόμαστε, διότι παρουσιάζει ελλείψεις και κενά η Ευρωζώνη ε, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά με το ότι είναι μια νομισματική ένωση χωρίς μια ε, οικονομική ένωση στην αγορά στην οικονομία της αγοράς. Θα συνεργαστούμε και με τους πράσινους. Σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι πρέπει να το εγκρίνουμε αυτά τα κείμενα και ως δικό μας, όχι μόνο άλλων. Εάν δεν αλλοιωθεί το περιεχόμενό του έτσι όπως έχει αυτή τη στιγμή. Φαίνεται ότι μερικές φορές έχουμε το εξής τικ. Πρέπει να βάλουμε τη λέξη διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις σε κάθε παράγραφο, αλλιώς δεν γίνεται. Είναι λίγο ψυχαναγκαστικό αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση ε, πρέπει να ολοκληρωθεί αυτό το οικοδόμημα της Ευρωζώνης. Ως εκ τούτου, συμφωνούμε με αυτούς τους τρεις πυλώνες, τη σύγκληση, την σταθερότητα και την επένδυση. Σύγκληση με κανόνες που μοιράζονται όλοι και που συμφωνούν όλοι, όχι σύγκληση με ε, το ε, τι κάνει κρόταφο. Δεύτερον, εργαλεία σταθεροποίησης των καταστάσεων ανισορροπίας και γι' αυτό γίνεται πρόταση για το επίδομα ανεργία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μένει να συζητηθεί, είναι ένα ενδεχόμενο, καλός. Το θέμα όμως είναι η πραγματική δημοσιονομική ικανότητα και η ικανότητα χρέωση, χρέωσης, δηλαδή σύναψης χρεών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα οποία ε, χρέη, δάνεια δηλαδή, θα αφιερωθούν στις επενδύσεις, επενδύσεις για να έχουμε αηφόρο ανάπτυξη, και για να απαντήσουμε σε αυτό που είναι το ζητούμενο σε κάθε ενιαίο οικονομικό χώρο που είναι η ενίσχυση αθρηστικά της ζήτησης. Θα έχουμε την ευκαιρία και να συζητήσουμε τις ε, τροπολογίες που έχουμε αφήσει κατά μέρος προσωρινά όταν συζητήσουμε την αντίστοιχη νομοθετική πρωτοβουλία και θα προσπαθήσουμε να έχουμε έναν οικονομικό χώρο στέρεο, δυνατό, που δεν θα είναι μόνο μια οικονομική βάση, αλλά σημείο κίνησης για την ανάκτηση της πολιτικής και κοινωνικής Ευρώπης, την οποία έχουμε αφήσει κατά μέρος μέχρι σήμερα. Ευχαριστώ. Κύριε Σεκχάτ. Ναι, ευχαριστώ πρόεδρε Θέμη. Σύντομο γιατί κάνουμε time sharing με τον συνάδελφο, όπως ξέρετε, το συνηθίζουμε. Όχι, όχι, εντάξει, δεν πειράζει. Αυτό που θα ήθελα να προσθέσω εγώ είναι το εξή, τα εξή δύο. Πρώτα, ευχαριστώ τους δύο συνεισηγητές που προβαίνουν σε αυτήν την πολιτική δήλωση, τοποθέτηση, γιατί περί αυτού πρόκειται και ξέρω ότι δεν ήταν καθόλου εύκολο να κερδίσουν την υποστήριξη των διαφορών πολιτικών ομάδων στο κείμενο που έχουν καταθέσει. Αν βάλεις ένα Γερμανό και μια Γαλλίδα μαζί, πάλι πάντα μπορείς να ξέρεις ότι θα υπάρχει αποτέλεσμα. Καλό είναι να βλέπουμε ότι υπάρχει αυτή η γαλλογερμανική συνεργασία πάντα. Αυτή ήταν η πρώτη παρατήρηση. Δεύτερον, αυτό που βλέπω εγώ ως πιο σημαντικό είναι το πολιτικό μήνυμα που στέλνουμε. Ότι το ευρώ όπως έχει τώρα χρειάζεται βελτίωση. Κατεπηγόντως. Η ιδέα ότι μπορούμε να αφήσουμε πίσω μας την κρίση του ευρώ και ότι όλα πάνε καλά, αυτή η ιδέα δεν υπάρχει και νομίζω ότι είναι ένα μήνυμα σαφέστατο από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και χαίρομαι που είναι σαφές αυτό το μήνυμα. Ε, υπάρχουν πολλές εκφράσεις που εγώ δεν θα χρησιμοποιούσα. Οι διαρθωτικέ μεταρρυθμίσεις και όλα αυτά, τα... οι εποδοί αυτέ τι οποίε βλέπουμε να ακούγονται και να γράφονται συχνά. Ένα τελευταίο σημείο κρίσιμη σημασία είναι το ότι αυτή η συζήτηση γίνεται και σε επίπεδο εθνικών κοινοβουλίων. Κάποιο παίζει μουσική από προεκλογική εκστρατεία, τουλάχιστον έτσι φαίνεται. Λοιπόν, ναι, είναι καλό να γίνονται αυτέ οι συζητήσεις και στα εθνικά κοινοβούλια, γιατί μπορούμε να κάνουμε μια σπουδαία συζήτηση για την αναγκαιότητα για δημοσιονομικό δυναμικό που τώρα βέβαια αυτή η συζήτηση γίνεται μια Τετάρτη βράδυ, αργά, κοντεύει 8 και είναι άδεια η αίθουσα. Αυτή η συζήτηση λοιπόν πρέπει να γίνει στα Εθνικά Κοινοβούλια. Και έτσι ξεκινάμε καλά. Τουλάχιστον έχουμε ένα σημείο κίνηση για τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ. Δεν βλέπω σαν συναλφό από το ομάδα EFTD, ούτε από το ENF. Προχωρώ λοιπόν στη διαδικασία ΚΑΡΣΤΙΑΕ. ο κύριος Χόκμαρκ, μετά ο κύριος Φερνάνδες. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ τους εισηγητές για το γαλλογερμανικό άξονα. Θα ήθελα να πω με κάθε μετριοφροσύνη ότι το σύμφωνο σταθερότητας η Γαλλία και η Γερμανία το υπονόμευσαν και και το δημοσιονομικό δυναμικό που θα έπρεπε αυτό να έχει. Και είναι σημαντικό αυτό γιατί είναι η ουσία της συζήτησης. Ε, ε ακούστηκε και ο Κέινς. Δεν θέλω να υπενθυμίσω στους φίλους όταν έγραψε ο Κέινς ε, τις θεωρίες του. Είναι πολύ πολύ πολύ παλιά. Και έχει εντωμεταξύ αποβιώσει ο Κέινς. Στα δε κράτη, στα οποία εφαρμόστηκαν οι ιδέες του, για να καταπολεμηθούν τα προβλήματα με μεγαλύτερα ελλείμματα, τα ελλείμματα μόνο μεγάλωναν και η ανταγωνιστικότητα μόνο μειωνόταν. Και θέλω για το γερμανό φίλο να πω ότι αυτό που πραγματικά εννοούσε ο Κέινς ήταν το σύμφωνο σταθερότητας. Γιατί ένα πλεόνασμα 3% και έλλειμμα 3% είναι το όνειρο κάθε καθηγητή οικονομικών, κάθε πανεπιστημιακού, όπως ο Κέινς. Αλλά δεν μπορέσαμε ποτέ στην πραγματικότητα να το τηρήσουμε αυτό. Εγώ λοιπόν που προέρχομαι από χώρα εκτός της ζώνης του ευρώ και θα ήθελα να μπούμε στην ευρωζώνη, πρέπει να πω ότι με καταπλήσει το γεγονός ότι η Σουηδία είναι μια από τι λίγε χώρες που εκπληρούν τα κριτήρια του ευρώ. Αυτό που έχω λοιπόν να, να πω είναι ναι, εμείς περάσαμε από κρίση, αλλά διδαχθήκαμε και είπαμε ότι θα πρέπει και οι θεσμοί να συνοδεύονται από πολιτικές. Δεν μπορεί καν να στηρίζεται μόνο σε θεσμούς, ούτε μόνο σε πολιτικές. Χρειάζεται να σέβεται και τα δύο. Και αυτά ε, θέλω να επισημάνω, γιατί δεν χρειάζεται να, να αυξήσουμε την ευρωπαϊκή φορολογία και τις δημόσιες δαπάνες, που θα ήταν μια συνέπεια αυτής της πρότασης γιατί έτσι θα υπονομευόταν η δημοσιονομική σταθερότητα, αλλά και η ανταγωνιστικότητά μας. Δεύτερον, το Ταμείο για τα Πρόβλεπτα. Θα ενημερώσω τους καλούς φίλους εδώ ότι η αδίποτε χώρα έχει πρόβλημα, θα μας δηλώνει όπως είναι απρόβλεπτο το πρόβλημά της. Και θυμάμαι ότι πριν από δύο-τρεις εβδομάδες που συζητούσαμε πάλι εδώ, εάν θα πρέπει να που κλείνουμε από το Σύμφωνο Σταθερότητας για τις χώρες της Ιβηρικής. Και όλοι είχαν ταχθεί κατά τη στήριξη των κανόνων. Άπαντες, πλην ορισμένων ολίγων. Θα ήθελα λοιπόν να πω κύριε Πρόεδρε ότι δεν πρέπει να λησμονούμε πως έχουμε δημοσιονομική δυνατότητα στο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να είναι ένα σταθερό και βιώσιμο σύμφωνο σταθερότητας και υπάρχει αυτό ο μπούσουλα στο Σύμφωνο σταθερότητα και ανάπτυξη, που δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε ούτε και μπορούμε να το αντικαταστήσουμε με νέους κανόνες. Ούτε μπορούμε να πούμε ότι δεν τηρούμε τους κανόνες και έτσι φτιάχνουμε καινούριου. Γιατί έτσι απλώς παραγνωρίζουμε τα πραγματικά προβλήματα της δημοσιονομικής δυνατότητας που είναι η ανταγωνιστικότητα και η ανάπτυξη. Και έτσι για να καταλήξω με τα συγχαρητήρια πάντα προς τους εισηγητές και τους και εισηγητές, θεωρώ ότι αυτή δεν είναι η λύση να δεν είναι η διέξοδος από τα ευρωπαϊκά προβλήματα. Σας ευχαριστώ. Είχε και επιφανέστατο οικονομολόγο τον κύριο Μίρνταλ η χώρα σας. Δεν ξέρω αν θα συμφωνούσε με σας. Δεν ξέρω αν θα διαφωνούσε μαζί μου ο Μίρνταλ, ο κύριος Χόκμαρκ, Πάντως όχι σήμερα. Καλύτερα να, κανείς ασαφώς, να, έχει κανείς ασαφώς δίκαιο παρά ε, συγκεκριμένα άδικο. Αλλά, εν πάση ο κύριος Φερνάνδες. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, θα μιλήσω γαλλικά. Νομίζω πως είναι η στιγμή, ακόμα και σε αυτή την αίθουσα βλέπω, πως η λέξη εμπιστοσύνη δεν υπάρχει. Και πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη καταρχάς ανάμεσα στα κρατημέλη. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει να μεταρρυθμίσουμε αυτή τη ζώνη. Υπάρχουν χώρες που κάνουν προσπάθειες ε, και άλλες που δεν κάνουν, που δεν έχουν εμπιστοσύνη γιατί πιστεύουν πως αυτές οι χώρες δεν κάνουν ε, ε, προσπάθειες, δεν σέβονται τους κανόνες, αλλά το πρώτο που χρειαζόμαστε είναι αυτή η λέξη εμπιστοσύνη που σε αυτή τη φάση δεν υπάρχει ανάμεσά μας. Και χρειάζεται η εμπιστοσύνη, όπως είπα, ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Πιστεύω και είναι η στιγμή να δώσουμε ένα μήνυμα. Αν όλα πάνε καλά, τα αφήνουμε. Όταν όμως υπάρχει πρόβλημα, κάτι που δεν λειτουργεί, τότε κάτι πρέπει να κάνουμε. Και θα έπρεπε να θέσουμε το ερώτημα γιατί υπάρχουν κανόνες που δεν γίνονται ποτέ σεβαστοί. Ο κανόνας του 60% του χρέους, ποιος το σέβεται. Το ΑΕΠ μάλλον για χρέος, ποιος το σέβεται. Ε, υπάρχουν κανόνες πρέπει να τηρούνται. Δεν πρέπει να ξεχνάμε και ότι εδώ δεν μιλάμε για κανονισμό. Είναι μια έκθεση πρωτοβουλίας. Σε μια έκθεση πρωτοβουλίας δεν χρειάζεται να πούμε πώς θα λειτουργήσει η παραμικρή λεπτομέρεια και πώς θα χρηματοδοτηθεί. Το ξέρουμε. Το Κοινοβούλιο δεν έχει καν την αρμοδιότητα να μιλήσει για τους ίδιους πόρους. Συμφωνώ με τη δομή. Όλα αυτά έχουν, ε, ε, αυτή η έκθεση έχει μέγα κύρος γιατί οι δύο εισηγητές έκαναν εξαιρετικό έργο για το οποίο τους ευχαριστώ. Συμφωνώ επίσης ε, ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε προς αυτή τη δομή με αυτούς τους πυλώνες. Ίσως να υπάρχουν διαφορές στο περιεχόμενο του κάθε πυλώνα, αλλά όμως συμφωνούμε για τους πυλώνες, πρέπει τώρα να δούμε το περιεχόμενο. Και υπάρχει κάτι που είναι σαφές, ότι μιλάμε πολύ αλλά στην πράξη δεν τα βάζουμε όλα αυτά. Είναι δηλαδή η ε, λυγική και ευθύνη. Και όταν μιλάμε για ευθύνη πρέπει να ε, σημαίνει ότι πρέπει να αποφύγουμε το moral hazard. Όταν μιλάμε για ευθύνη, υπευθυνότητα σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχουν όροι. Πρόκειται για τον σεβασμό των κανόνων. Χρειάζεται περισσότερη διαφάνεια, περισσότερη νομιμοποίηση, περισσότερη δημοκρατία. Καλύτερη διακυβέρνηση. Πιστεύω επίσης πως υπάρχουν άνθρωποι που είναι κατά το ευρώ και που θα είναι πάντα κατά μιας έκθεσης, ό,τι και αν γίνει. Αλλά αυτοί που επιθυμούν την αλληλεγγύη την πιθανότητα, μια ε, δυνατότητα πρόβλεψης και μέσα για την ανάκτηση θα πρέπει να συμφωνήσουμε και θα ήταν κακό να δώσουμε τέτοιο μήνυμα ότι για μας, για το Ευρωκοινοβούλιο όλα πάνε καλά και το μόνο πρόβλημα που, έχουμε, που χρειαζόμαστε μάλλον είναι να σεβαστούμε αυτά που υπάρχουν αλλά που κανείς δεν τα, δεν τα σέβεται. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω άλλο να μιλητεί στον καταλογό μου, οπότε θα κάνω κι εγώ μια σύντομη παρέμβαση, γιατί μπαίνω στον πειρασμό με, με αυτά που είπε ο κύριος Χόκομαρκ. Γιατί πρέπει να πω ότι σε αυτή την έκθεση δεν βρίσκω καθοδήγηση για την εφαρμογή του, του Συμφώνου Σταθερότητας. Δεν δεν είναι κενσιανή λογική, ούτε μη κενσιανή. Αντιμετωπίζει διαφορετικά το θέμα. Το γεγονός ότι δεν έχουμε δυνατότητα σταθεροποίησης σε επίπεδο ευρωζώνης, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να εξαρτώμεθα από την νομισματική πολιτική και από τους εθνικούς προπολογισμού από την άλλη πλευρά, που μπορεί να δημιουργήσει ακριβώ το πρόβλημα τη υπερβολική στηρίξη στο, στο στην νομισματική πολιτική, γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα απορρόφησης του, του σοκ και θα πρέπει να κόψουμε τις επενδύσεις γιατί δεν έχουμε λειτουργία ασυμμετρικής απορρόφησης του, των σοκ και πρέπει μετά να βασιστεί στον εθνικό προπολογισμό για να κάνεις κάτι το οποίο όμως δεν μπορεί να το κάνει ο εθνικός προπολογισμό. Προσωπικά λοιπόν βρίσκω την ιδέα μιας ε, δημοσιονομικής δυνατότητας συνεπή με την άποψη ότι χρειάζεται πλήρως ισορροπημένος προπολογισμό σε εθνικό επίπεδο και αυτό μπορείς να, κάνεις, να το κάνεις αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα για σταθεροποίηση και απορρόφηση. Διαφορετικά πρέπει να υπάρχει αυτή η δυνατότητα και αυτή η λειτουργία. Το δουνουτού επίσης είναι σαφές. Είναι μια τεχνική ανάλυση και δεν έχει να κάνει το να απορροφήσει τα συμμετρικά σοκ με το αν έχει ε, δημοσιονομική πολιτική επεκτατική ή λιγότερο επεκτατική. Μπορεί να έχει διαφορετικές απόψεις για τη δημοσιονομική πολιτική όσον αφορά τον κύκλο, αλλά είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Δεν θα ήθελα λοιπόν να μετατραπεί αυτή η συζήτηση σε μια συζήτηση όπου χρειάζεται, για το αν χρειάζεται ή όχι να σεβαστούμε την δημοσιονομική πολιτική. Όχι, δεν είναι αυτός ο στόχος της έκθεσης. Ο στόχος της έκθεσης είναι να δούμε αν η Ευρώπη χρειάζεται επίσης πέρα από τους δύο πυλώνες της εθνικής ε, δημοσιονομικής πολιτικής και της κοινή νομισματικής πολιτικής να φτιάξει και μια λειτουργία, μια κοινή λειτουργία. Πρώτον για να την, την μεταρρύθμιση και είναι, μπορεί να αντιμετωπίσει τα ασυμμετρικά σοκ αλλά και τα συμμετρικά. Ε, μπορούμε, μπορεί να διαφωνήσουμε για την δημοσιονομική πολιτική στην έκθεσή μας στην ετήσια για το IDS που, που επίσης βρίσκουμε ε, συμβιβαστικέ και ισορροπημένη προσέγγιση. Οπότε αυτή η έκθεση να μην τη φορτώσουμε με πράγματα τα οποία δεν είναι εντό θέματο. Έπειτα για το θέμα του Υπουργού Οικονομίας και αυτό συνδέεται εδώ αυτό, γι' αυτό θέλω να είμαι πιο σαφής και αστιεύτηκα για να ξεκινήσω από τα όσα είπε ο κύριος Μόρεσαν, Ακριβώς για να ακολουθήσουμε και την λογική του κύριου Τάγκο, ότι δηλαδή το να έχουμε την καλύτερη δυνατότητα για να διακρίνουμε ε, ευρωπαϊκές και εθνικές αρμοδιότητες, οικοδομώντας σταδιακά μια δημοσιονομική δυνατότητα που μπορεί να καταλήξει στη, στον Υπουργό Οικονομίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι βάζουμε άλλο ένα ακόμα στοιχείο διζητικότητας ή διαχείρισης ε, της δημοσιονομικής πολιτικής σε εθνικό επίπεδο. Όχι. Αντίθετα θέλουμε να μπορούμε να διακρίνουμε και να βρούμε και περισσότερους αυτοματισμούς ή πειθαρχία της αγοράς ή ίσως και δυνατότητα ε, αποτυχίας του εθνικού προϋπολογισμού. Αυτά είναι συμβατά. Και γι' αυτό ακριβώς είμαι βέβαιος ότι θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε σε μια κοινή βάση που είναι αυτό το έγγραφο που είναι μια πολύ σημαντική συμβολή του Κοινοβουλίου στην στήριξη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και αυτό βέβαια δεν σημαίνει τίποτα για το ποια άποψη μπορεί να έχει κάθε πολιτική ομάδα για την δημοσιονομική πολιτική. Αυτό είναι ένα διαφορετικό θέμα. Δεν είναι αυτό το θέμα του της έκθεσης. Ζητώ συγγνώμη για αυτή ε, μου την παρέμβαση και το... θέλετε μάλιστα ο κύριος Χόκμαρκα. Ναι, καταρχάς ε, με τιμά που οι ταπεινές μου παρατηρήσεις ε, προκάλεσαν αυτήν την συζήτηση τόσο αργά εγώ θέλω να πω τι είναι ε, τα συμμετρικά σοκ και η χαλεπή καιρή. Τι είναι η χαλεπή καιρή, είναι πάντα θέμα ε, ορισμού και έχω μάθει το εξής. Τα συμμετρικά σοκ είναι αυτά που σε χτυπούν εσένα και τα αυτά που χτυπούν τους άλλους μπορεί να είναι συμμετρικά. Ε, δεύτερον, εάν έχεις μία, μία αποδοτική οικονομία για χρόνο, για καιρό, θα το λέμε πάντα ότι είναι χαλεπή καιρή παρότι μπορεί αυτό να οφείλεται στην οικονομική σου πολιτική ή στις υπερβολικές δαπάνες. Γι' αυτό αυτά τα δύο συνδέονται. Στην πραγματικότητα, η βασική, η βασική δημοσιονομική δυνατότητα στην πραγματικοτητα η βασικη βασικη δημοσιονομικη δυνατοτητα στην ενωση θα πρέπει να είναι στα κράτη-μέλη και πρέπει αυτά να διαχειρίζονται σωστά. Και το βασικό πρόβλημα που έχουμε τώρα με τη δημοσιονομική δυνατότητα είναι ότι δεν υπάρχει σωστή διαχείριση. Και το να φτιάξουμε ακόμα μια δημοσιονομική δυνατότητα εμέσως θεωρεί ότι δεν θα ακολουθήσουμε τους κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας. Αυτό θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από ό,τι θα λύσει, κατά τη γνώμη μου. Τότε όμως μπορεί να μην χρειαζόμαστε, αν ακολουθήσουμε αυτή τη λογική, ούτε καν τον προϋπολογισμό της Ένωσης. Ε, να δώσω το λόγο πάλι στους συζητητές για να κλείσουμε. Ευχαριστώ. Είναι αργά, αλλά έχουμε φτάσει στην ουσία της συζήτησης. Ε, κρίμα που δεν ήσασταν εσείς οι σκιώδες εισηγητής. Θα μπορούσατε να είχατε θέσει αυτά τα ζητήματα νωρίτερα. Όμως, αφού τέθηκαν τα ζητήματα από τους μεν και τους δε, να πω και εγώ δύο πραγματάκια που οδήγησαν στη σύνταξη αυτής της έκθεσης. Όταν υιοθετήσαμε το ευρώ, συμφωνήσαμε πάνω σε συγκεκριμένους ε, κανόνες που δεν τηρούνταν αρκετά. Και με την πάροδο των ετών προσπαθήσαμε να συμπληρώσουμε τους κανόνες, να τους τελειοποιήσουμε και κάποια στιγμή προ... υπήρξε πρόσκρουση σε αυτό το θέμα της ιδιοκτησίας από τα κράτη-μέλη. Πέσαμε πάνω σε αυτό. Και αντί να χτυπάμε το κεφάλι μας στον τοίχο, τείχος όντας η εθνική κυριαρχία των κρατών μελών και η άσκηση οικονομικής πολιτικής από αυτά, και κανείς δεν τον αμφισβητεί αυτό, είπαμε να έχουμε ένα κώδικα σύγκλησης, έτσι ώστε τα κράτη-μέλη σιγά σιγά να μεθούν έντονα και αρκετά για τις δικές τους στρατηγικές οικονομικής πολιτικής χωρίς να έχουν την αίσθηση ότι ε, θα δρούν επειδή θα τους διατάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και ε, κάτι τέτοιο θα ήταν ούτως ή άλλως αντιπαραγωγικό και όχι οδηγός για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των κρατών μελών. Αυτό καταρχάς. Κατά δεύτερο, ως προς τα ασύμετρα σοκ, είπε ο προηγούμενος ομιλητής ότι δεν ξέρουμε τι είναι αυτό. Εν πάση περιπτώσει αυτό που ξέρουμε είναι ότι μετά την υιοθέτηση του κοινού νομίσματος πρέπει να ξαναδιαβάσουμε ε, το βασικό εγχειρίδιο της οικονομικής επιστήμης. Έστω, ο Κέινς δεν είναι πια στη μόδα, αλλά αν εξετάζει κανείς τη λειτουργία της ζώνης του ευρώ, ε, δεν απαγορεύεται ε, να δούμε τι είχαν πει οι ιδρυτές πατέρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την έκθεση Μακντούγκαλ ε, μεταξύ άλλων, όπου ε, τα περιεχόμενα αυτά της έκθεσης τότε δεν, δεν έχουν ληφθεί υπόψη, ποτέ δεν ελήφθησαν υπόψη. Έχει φύγει, έχει φύγει ο κύριος Χόκμαρ, ίσως πρέπει εδώ να σταματήσω να του απαντάω. Όμως, σε κάθε περίπτωση Σαφέστατα, ο δικός χάρτης λέει ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να βασιστούν στις δικές τους δυνάμεις, πρέπει να καταβάλουν τις δικές τους προσπάθειες για να ε, διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Δεν μπορούμε όμως να συνεχίσουμε μια κατάσταση κατά την οποία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε επίπεδο ζώνης του ευρώ δεν υπάρχουν εργαλεία για την αντιμετώπιση των σοκ που υφίσταται μια οικονομία είτε είναι ασυμμετρικά είτε είναι συμμετρικά αυτά τα σοκ. Κάθε οικονομία διαθέτει τέτοιου είδους εργαλεία και στην ευρωζώνη δεν έχουμε μπορέσει να το υλοποιήσουμε μέχρι σήμερα παρά μόνο σε συνθήκες κρίσης και μάλιστα ατελώς έγινε επίκληση στον Κέινς. Υπόθηκε ότι δεν είναι πια της μόδας. η ακραίως φιλελεύθεροι είναι σήμερα της μόδας, αναρωτιέμαι. Εάν δούμε τον απολογισμό των ετών Ρίγκαν και Θάτσερ, δεν είναι η στιγμή, πιστεύω, να εμφορούμαστε από δόγματα και να τα αντιπαραβάλλουμε μεν, με τους δε. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να διασφαλίσουμε ότι το ευρώ μπορεί να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των κρατών που μοιράζονται αυτό το κοινό νόμισμα. Και γι' αυτό, ό,τι προτείνουμε σε αυτόν τον δικό χάρτη θα πρέπει να το ακούσει και να το λάβει υπόψη της Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τη σύνταξη της Λευκής Βίβλου, όπως επίσης το ίδιο οφείλει να πράξει και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν θα αντισταθώ στον πειρασμό να απαντήσω σε ένα επιχείρημα των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών. Ότι δηλαδή με αυτό τον οδικό χάρτη μειώνουμε την εθνική κυριαρχία των κρατών μελών. Αντιθέτως πιστεύω, όλη αυτή η ιδέα του κώδικα σύγκλησης επιτρέπει στα κράτη-μέλη να ανακτήσουν το περιθώριο ελιγμών ε, σε ό,τι έχει να κάνει με τις οικονομικές πολιτικές τους και σε κάθε περίπτωση επιθυμώ να έχουμε τη μέγιστη δυνατή συνένεση, ε, μια στέρεα πλειοψηφία για να μπορέσουμε να στείλουμε αυτό το ηχηρό πολιτικό μήνυμα. Ο κύριος Μπέγκε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Yeah. Ναι. Συμπλήρωσαν και βλέπω να αποχωρεί ο συνάδελφος. Στα όσα είπε για, την, ε, για το ownership, την ιδιοκτησία, την αποδοχή. Ε, θα το καταφέρουμε αυτό μόνο εάν μπορέσουμε αφενός με να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη ευθύνη, υπευθυνότητα για το συμβαίνουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διακυβέρνηση και λογοδοσία για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και για τα εθνικά αντίστοιχα που χρειάζεται να βελτιωθούν η λογοδοσία και η υπευθυνότητα και η διακυβέρνηση κατεπηγόντως αλλά ταυτόχρονα και με αυτά που έχουμε δει από τις οικονομικές υπηρεσίες και τα, οι συστάσεις ανακράτους που έχουμε εξετάσει εδώ στο Κοινοβούλιο και τη διημόρφωση αυτών των συστάσεων στα κράτη-μέλη έχουμε διαπιστώσει το εξής ότι γίνεται πάρα πολλή δουλειά στα κράτη-μέλη με πολλές, πολλούς πίνακες με θετικά στοιχεία σε ορισμένε σε κάποια άλλη όμω όχι. Και πια εκεί αρχίζει η ουσία, διαφάνεια και λογοδοσία. Και χρειάζεται ένα μηχανισμό που έχει και σήμερα και σε άλλε περιστάσει αναφερθεί. Ένας μηχανισμός που σημαίνει περισσότερη επαγγελματικότητα, έτσι ώστε να μπορέσουμε εμείς, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια, να συνεργαστούμε και να μην είμαστε σε μια διαρκή αντιπαράθεση. Αλλά να καταλήξουμε επιτέλους σε αυτό που θα μπορούσα να περιγράψω ως ευρωπαϊκή κοινή γνώμη που δεν υπάρχει ακόμα. Νομίζω ότι μόνο με καλή συνεργασία μεταξύ μας μπορούμε να καταλήξουμε σε καλές θέσεις και λύσεις. Τοποθετήθηκαν επικριτικά κάποιοι συνάδελφοι απέναντι στην ε, πρότασή μας. Το λαμβάνουμε υπόψη, να ακούσαμε με προσοχή τις παρατηρήσεις τους. Θέλω να επισημάνω πάντως ότι έχουμε κάνει σημαντική προσπάθεια αυτές τις βασικές θέσεις να τις ενσωματώσουμε στο κείμενό μας. Και τώρα πια έχει έρθει η ώρα να προχωρήσουμε σε ουσιαστική βελτίωση του τελικού κειμένου για την ανάπτυξη της, του δυναμικού, του μεσονομικού δυναμικού. Αυτά έχουμε να προσφέρουμε, αυτά έχουμε να προσθέσουμε. Και σημειώνω ότι δεν θα πρέπει να ανατραπούν οι ισορροπίες αυτού του δικού χάρτη. Πρέπει να παραμείνει μια ισορροπία που θα είναι αποδεκτή από τις ομάδες. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος, σύντομη και χρήσιμη η συζήτηση. Έχετε κάτι να προσθέσετε κύριε συνάδελφε. Όχι. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε και τα επόμενα βήματα. Περιμένουμε τα επόμενα βήματα λοιπόν για αυτή τη σημαντική ελπίζουμε συμβολή στην ΟΝΕ.